Πρώτη ε, έκθεση είναι η έκθεση Γάουτα. όσον αφορά πρωτόκολλα για θέματα ειδικά ε, του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. διονομαστικής κλήσεως ε, η ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία. Έκθεση Σβόμποντα. Σύμβαση της Χάγης της 30 Ιουνίου 2005 σχετικά με συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας. ονομαστική κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε στην έκθεση Σαρβαμά. Κινητοποίηση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Votazione Πέρα της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση για τενμάκι, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι το κεφάλαιο που αφορά τη Γαλλία, διονομαστικής κλίσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Πέρας. Εγκρίνεται. Φτάνουμε σε αίτημα γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις συνθήκες συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων από τις ε, καταστάσεις επιβατών PNR. Το λόγο έχει ο κύριος Μπροκ. Κύριε Μπροκ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εξ ονόματος ε, της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, θέλω να ζητήσω ε, αναβολή του ψηφίσματος αυτό για το Δεκέμβριο δυνάμει του άρθρου 190 ε, εδάφιο 4 του κανονισμού. Παρακαλώ την ε, Επιτροπή που το ζήτησε ε, τη ΛΥΜΠΕ να το καταλάβει ε, έχει επιπτώσεις διότι μια γνωμοδότηση, ένα προδικαστικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 30 μήνες. Ο παράγων χρόνος είναι κρίσιμος ε, πολιτικός παράγων σε τέτοια σημαντικά θέματα. Παρακαλώ να συμμετέχουν η ΛΥΜΠΕ, η ΑΦΕΤ, όλες οι αρμόδιες επιτροπές για να δούμε πραγματικά τι συνέπειες θα έχει ένα τέτοιο ερώτημα προς το δικαστήριο. Παρακαλώ να βληθεί για τον Δεκέμβριο και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Υπήρξατε σαφέστατος. Ένας ε, ομιλητής υπέρ, ε, ένας ομιλητής ο οποίος θα είναι υπέρ της προτάσεως του κυρίου Μπρόκ. Παρακαλώ. Oh, ο κύριος Φως. Φως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω με χαρά την πρόταση αυτή, διότι αυτή η διαδικασία δεν ε, ήταν κάτι που είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους οι σκιώδη ηγητές, ούτε στην ομάδα μας είχαμε αρκετό χρόνο να σκεφτούμε την εμβέλεια και τις συνέπειες όλων αυτών και να τις συζητήσουμε και το θεωρώ ε, σκόπιμο να το συζητήσουμε γιατί όλοι θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει, τι συνέπειες θα έχει ε, για τις εταιρικέ μας σχέσεις με άλλες χώρες, για τις αεροπορικές εταιρείες και την πολιτική μας ευθύνη. Διότι εμείς είμαστε ο νομοθέτης και όχι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πρέπει καμιά φορά να αρχίζουμε να αναλαμβάνουμε και πολιτικές ευθύνες εδώ μέσα. Ευχαριστώ κύριε Φως. Τώρα ε, ένας ομιλητής ο οποίος θα αντιτίθεται σε αυτή την πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Παραλίγο να πω, πω, πω, τι γλυκά είναι αυτά που μας λέτε. Τις τελευταίες ημέρες άκουγα πάντα ότι μια διαδικασία ενώπιον του δικαστηριού μπορεί να χρειαστεί ε, μέχρι και δύο χρόνια από τους αντιπάλους. Τώρα τα δύο χρόνια έγιναν 30 μήνες. Αν συζητήσουμε άλλη μια εβδομάδα μπορεί να πάνε και τέσσερα χρόνια. Ε, κατά τα άλλα, ε, θέλω να θυμίσω ότι ο Πάπας μόλις ε, μας είπε ότι... ότι πρέπει να δεχόμαστε τους ίδιους μας τους κανόνες και τις αξίες. Και εγώ τον άκουσα. Και εσάς άκουσα. Και τώρα, είτε ψηφίσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, είτε είναι αποτέλεσμα εκλογών, μπορεί και τα δύο να μην σας αρέσουν. Ε, ωστόσο, θα πρέπει ένα αποτέλεσμα ψηφοφορίας να το σεβόμαστε και να το δεχόμαστε. Εχθές ψηφίσαμε, ήταν σαφές το αποτέλεσμα και τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτή την απόφαση για το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ευχαριστώ κυρία Επομένως θα ψηφίσουμε το αίτημα το οποίο υπευλήθη διανατάσεως της χειρός υπέρ της αναβολής κατά είναι απαραίτητο να γίνει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. E Περνάμε λοιπόν ε, στην ψήφιση του ψηφίσματος. Διονομαστικής κλίσεως επί του συνόλου του ψηφίσματος άρχεται. Votazione chiusa. Πέρας της ψηφοφορίας. Περνάμε τώρα στην έκθεση STEER. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Παγκόσμιο Πλαίσιο Ανάπτυξης για την ε, περίοδο μετά το 2015. Παράγραφος 4. Ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση όπως θέλετε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Και η παράγραφος 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22 σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα Άρχεται η ψηφοφορία πάντα διονομαστικής κλίσεως. Παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Τρίτο τμήμα. Διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Τέταρτο τμήμα διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση βεβαίως άρχεται Votazione Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 32 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Πρώτο τμήμα της παραγράφου 37. Υπέρ. Approvato. Seconda parte. Δεύτερο τμήμα διανομαστικής κλήσεως άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 58 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση θέλετε πολύ ωραία άρχεται πέρας εγκρίνεται Περνάμε στην παράγραφο 61 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 68 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διονομαστικής κλίσεω άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πάντα διονομαστικής κλίσεω άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 74. διατάσεις της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Ποτατσιόνι Πέρας. Εγκρίνεται η παράγραφος 74. Παράγραφος 78, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διανατάσεως ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Παράγραφος 78, τμήμα 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. αιτιολογική σκέψη ο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του, διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Στυρ. Περνάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, παράγραφος 1, διανατάσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται Votazione chiusa. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Διανατάσσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα πάντα διονομαστικής κλίσεως ε, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30 σε δύο τμήματα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32 διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 35, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Παράγραφος 40, τροπολογία 1, διονομαστικής κλίσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 45 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Πέρας. Approvato. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 46, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ψηφίζουμε στο σύνολό του το ψήφισμα διανατάσεως της χειρός υπέρ κατά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 επεξηγήσεις ε, ψήφου. Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν, παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα και τους εύχομαι ε, καλή όρεξη. Συνεχίζουμε εμείς τη συνεδρίασή μας.